εκθέσεων σύντομα ξεκινώντας από την έκθεση της ε, κυρίας Λούνατσεκ με θέμα ομοφοβία και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Και πρώτα θέλω να παρακαλέσω την ε, εισηγήτρια να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Δεν περίμενα τόσο μεγάλο αριθμό ε, μηνυμάτων στο ε, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πάνω από 40.000 που λένε όχι στην έκθεση Λούνατσεκ. Μάλιστα ε, κάποιοι hackers επιτέθηκαν και στην προσωπική μου ιστοσελίδα. Δεν ξέρω ποιος ήταν, ε, μπορεί να είναι σύμπτωση, μπορεί και όχι. Τέτοια αντίδραση σε μια έκθεση που κατά βάση τι κάνει, μιλάει για τα δικαιώματα των ανθρώπων να αγαπούν και να ζουν τη ζωή τους χωρίς φόβο. Δεν περίμενα τέτοια αντίδραση. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να ξεκινήσω την ε, παρουσίαση της έκθεσής μου ε, απευθυνόμενη σε, κυρίως σε ε, όσους και όσοι από εσά νιώθουν τα ίδια αισθήματα αντίδρασης από την έκθεση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, θα θέλατε η κόρη σας ή ο γιος σας ο αδελφός σας ή η αδελφή σας να φοβάται, να ε, περπατάει χέρι με χέρι με τον αγαπημένο του ή τον αγαπημένο της ε, στους δρόμους. Θα θέλατε να φοβούνται ε, τη Δευτέρα το πρωί να πούνε στους συναδέλφους στο γραφείο με ποιον πήγαν σινεμά Κυριακή βράδυ ή θα θέλατε ένας φίλος σας να φοβάται να σας πει ότι ε, έχει ερωτευτεί έναν άντρα ή μια φίλη σας ότι έχει ερωτευτεί με μια γυναίκα. Φαντάζομαι πως όχι. Φαντάζομαι πως θα λέγατε σε αυτούς τους ε, φίλους ε, να σας μιλήσουν, ε, να σας εξηγήσουν γιατί νιώθουν φόβο. Ε, γι' αυτό αυτό αφορά η έκθεση. Θέλω να εξασφαλίσουμε ότι οι λεσβίες και οι ομοφιλόφιλοι, καθώς επίσης και οι αμφιφιλόφιλοι, διαμφιλικοί και διαφιλικοί, θα μπορέσουν να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς διακρίσεις εναντίον τους, χωρίς φόβο, με και να ε, τους συμπεριφέρονται με σεβασμό στην ιδιωτική και τη δημόσια ζωή τους ε, ως πολίτες αυτής της κοινή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μιλούμε για κάποια ιδιαίτερα δικαιώματα, όπως λένε ορισμένοι στα email που μας στείλανε. Όχι. Δεν πρόκειται για ιδιαίτερα δικαιώματα. Ε, δεν ζητούμε ιδιαίτερα δικαιώματα. Ούτε προνόμια. Θα ήθελα να μου πείτε ένα, ένα μόνο ειδικό δικαίωμα που αναφέρει η έκθεσή μου, που θα έδινε ένα προνόμιο στους ΛΟΑΔ. Ένα δικαίωμα το οποίο άλλοι εναντίον των οποίων υπάρχουν διακρίσεις, Ρωμά κλπ. δεν διαθέτουν και δεν μπορούν να ασκήσουν. Το δικαίωμα να, πάνε, να πηγαίνουν σε σχολεία χωρίς να τους εκφοβίζουν. Το δικαίωμα να μην θεωρούνται ψυχικά ασθενείς. Το δικαίωμα να μην απολύονται από τη δουλειά τους εξαιτία του με ποιον ε, μοιράζονται τη ζωή τους. Κυρίε και κύριοι, έχουμε στρατηγικές για να καταπολεμούμε τις διακρίσεις εναντίον των Ρωμά, για παράδειγμα, εναντίον των ανθρώπων με αναπηρίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη δέκα φορές έχει ζητήσει από τον Επίτροπο να υποβάλει οδικό χάρτη κατά της ομοφοδίβειας ε, και κατά των ατόμων ΛΟΑΔ. Δεν το έχει κάνει. Γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή Ελευθεριών, η Επιτροπή αποφάσισε να ε, ε, συντάξει αυτή τη γνωμοδότηση. Η, ε, η Υπηρεσία Θεμελιών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι 93.000, ότι σε μια, ε, το 60% από 93.000 άτομα ΛΟΑΤ που, που απάντησαν στην έρευνα φοβούνται. Ένας στους τέσσερις ε, έχει δεχθεί απειλές ή επιθέσεις τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό είναι η ομοφοβία. Και δεν είναι δυνατόν να το ανεχθούμε πλέον στην Ευρώπη. Πολλοί από εμά. ΛΟΑΔ. Έχουμε ζήσει τη ζωή μας μέσα στο φόβο για πολύ καιρό. Στην έκθεσή μου λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενεργήσει. Αυτό πώς θα γίνει. Όχι ε, υπερβαίνοντας τι αρμοδιότητές της. Ούτε εμπλεκόμενη με τι αρμοδιότητες των κρατών μελών. Το καθιστούμε σαφέ αυτό. Κοιτάξτε την παράγραφο 5. Θα πρέπει να προστατευτούν οι ε, αρμοδιότητε των ε, υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών. Όμω, κάτι πρέπει να κάνουμε. Η έκθεση λέει στην Κομισιόν, αυτή και την επόμενη Κομισιόν και λέει και σε εμά εν το μέσο της προεκλογικής εκστρατείας μας, ότι θα πρέπει να εργαστούμε για να καταπολεμήσουμε το φόβο, να εξασφαλίσουμε ότι όσοι διώκονται ε, ή εκφοβίζονται ε, εξαιτία του ότι είναι ομοφιλόφιλοι ή λεσβείες θα μπορούν να πάνε στην αστυνομία και οι αστυνομικοί θα, καταλαβα... θα καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επίσης ότι στα σχολεία, για παράδειγμα, ότι στα σχολεία θα ε, εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές. Θα γίνεται λόγος, θα μιλάνε στα, στους μαθητές ότι υπάρχουν οι ΛΟΑΔ και δεν είναι δυνατόν να υφίστανται αρνητική μεταχείριση. Ευχαριστώ. Very much. This is Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Πολλοί θέλουν να πάρουν το λόγο, όπως φαντάζεστε, στα πλαίσια του ΚΑΣΤΙΑΗ. Θα δώσω σε όλους το λόγο. Αλλά θα κλείσω εδώ τον κατάλογο. Η κυρία Ζαμπόσκα είναι η πρώτη. správa Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα το οποίο διχάζει την κοινή γνώμη. Η ψηφοφορία αύριο πιστεύω θα δείξει ότι και το Κοινοβούλιο διχάζεται. Εγώ θα υπερψηφίσω την τροπολογία υπαριθμών 1 αύριο που προτείνει ένα εναλλακτικό ψήφισμα. Αυτό θέλουν οι ψηφοφόροι μου και εγώ είμαι υπέρ της ε, αρχής των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσω να πείσω στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για την αποτελεσματική υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποστηρίξω την προστασία και επιβολή των ανθρωπινών δικαιωμάτων και την ισορροπία μεταξύ των επιλογών και του δικαιώματος της ζωής και άλλων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει η ΛΟΑΔ όχι να έχουν περισσότερα δικαιώματα, αλλά να είναι ίσοι Μπορεί να μην σα αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, η ΛΟΑ. Δεν έχει σημασία. Μια πολιτισμένη κοινωνία όμω κρίνεται από το πώ ε, αντιμετωπίζει τι μειονότητέ τη. Και 28 χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, πολλά ακόμα να κάνουν. Η αντίθεση σε αυτή την έκθεση αποδεικνύει ότι πρέπει να λάβουμε δράση για να καταπολεμήσουμε τι διακρίσει και το μίσος. Η μυσαλλοδοξία που υπάρχει είναι τρομερή ε, στον 21ο αιώνα. Γιατί δεν θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί, οι ΛΟΑΔ, να έχουν τα ίδια, τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους. Όχι προτιμησιακά δικαιώματα, ίσα δικαιώματα. Τελειώντας, πρώτα θέλω να πω το εξή. Ε, οι ψηφοφόροι μου θέλουν να είμαι θαραλέος και να κάνω το σωστό πράγμα. Θα υπερψηφίσω την έκθεση Λούνατσεκ, γιατί ως κοινωνία θέλουμε να αντιμετωπίζουμε όλους με τον ίδιο τρόπο και πολιτισμένα ή όχι και να μην πετάξουμε στα σκουπίδια όλα όσα κατάφεραν να, πετύχουμε, να πετύχουν γενιές επιγενεών. Bilbao. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα στηρίξω αυτό τον οδικό χάρτη για να προστατέψουμε θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των Ευρωπαίων που απειλούνται σήμερα. Ε, περίπου 50% του πληθυσμού των ΛΟΑΔ τον τελευταίο χρόνο ε, ήταν ε, θύμα απειλών και η μισή από αυτούς και βίας. Ε, η ελευθερία ε, του, η σεξουαλική ελευθερία είναι μία από τις ελευθερίες που πρέπει να προστατεύουμε. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ηγηθούν σε αυτόν τον αγώνα μια στιγμή που οι πιο συντηρητικές ε, δυνάμεις νοσταλγούν ε, το, την εποχή που ο κόσμος ΛΟΑΔ δεν υπήρχε. παρόλο που τους καταδίκαζαν σε φυλάκιση και περιθωριοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο, μάλιστα, ε, προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή μας από τα άλλα προβλήματα φτώχειας κλπ. Ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ελευθερία όλων. Ευχαριστώ. Εγώ, κύριε Μπιλμπάου. ο συνάδελφος Ήρα Ζαμπαλμπέτια. Χαίρομαι που έφτασε αυτή η έκθεση στην Ολομέλεια. Πρόκειται για μια πολύ καλή γνωμοδότηση που ελπίζω ότι θα βοηθήσει τον αγώνα κατά της ομοφοβίας ε, και, της, των διακρίσεων βάσει το σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα του φύλου. Ελπίζω ότι θα πιεστούν τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν αποτελεσματικές πολιτικές για αυτά τα θέματα σε σχέση με τους ΛΟΑΔ και υπέρ των δικαιωμάτων τους. Ελπίζω επίσης ότι ορισμένα κράτη-μέλη ε, θα σκεφτούν, κράτη-μέλη όπως η Πορτογαλία και η Κροατία, ε, όπου ε, έχουν, ε, παραβιάζονται τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ. Συγχαίρω την συνάδελφο Λούνα Τσέκ για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε point of order. Do you have a point of order, Ms. Morvai? Διαδικαστικό, κύριε Μορβάη. Sir, can you explain your point of order? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Φυσικά. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Η μπλε κάρτα. Τι κάνετε με την μπλε κάρτα. Τι, λέει, τι λένε οι κανόνες διαδικασίας. Γιατί εγώ ύψωσα την μπλε μου κάρτα ε, δύο, πριν μιλήσουν πριν δύο μιλητές. Με είδατε, οι βοηθοί σας με είδανε, αλλά με αγνοήσατε πλήρως. Να σας εξηγήσω. Το έχω ξαναεξηγήσει. Είπα ότι θα δεχθώ όλα τα αιτήματα λόγου για το Catch the Εν συνεχεία, αποφάσισα να μην δεχτώ τις μπλε κάρτες, ούτως ώστε να γίνει μια πολιτισμένη συζήτηση στην Ολομέλεια. Μπορείτε να ζητήσετε το λόγο στα πλαίσια διαδικασία Catch the Eye, αλλά όχι με την μπλε κάρτα. Δεν θα επιτρέψω καμία μπλε κάρτα σε αυτή τη συζήτηση. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλλον δεν θα είναι και η τελευταία φορά. Πολύ συχνά την πέμπτη το απόγευμα συζητάμε τι γίνεται σε άλλες χώρες, τη στάση που έχουν στη Ρωσία, την Αφρική, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ορθώς το συζητάμε. Πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουν τη ισότητα για όλους. Στα κράτη-μέλη και, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είπε και ο Μάικλ Κάσμαν. Πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους αυτούς. Εγώ είμαι φύλαφλος και χάρηκα πάρα πολύ που πολλοί ποδοσφαιριστές και αθλητές ε, και μάλιστα δρομής τεμποδίων βγήκαν και είπαν ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφιλοι. Πρέπει να δεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να δώσουμε και να εξασφαλίσουμε ισότητα, την ισότητα σε όλους. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ πολύ. Και Ουλρίκε, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη θαραλέα έκθεση, η οποία έρχεται αυτό το χρόνο αποδεικνύοντας δε, πόσο τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι ιδιαίτερα ειδικά δικαιώματα, είναι αυτά τα οποία ρυθμίζουν τη ζωή μας και μάλιστα επί τη βάση και τη αρχή ότι είναι όλοι άνθρωποι ίσοι. Ε, σε αυτό λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε και στην εξέλιξη του πολιτισμού της Ευρώπης με τη συζήτηση αυτή. Η έκθεση αυτή με βρίσκει σύμφωνη γιατί τάστε κατά της, των διακρίσεων εις βάρος των ανθρώπων που ζουν διαφορετικά από τους άλλους. Δύο άνδρες μαζί, δύο γυναίκες μαζί ή ενδεχομένως και με άλλη σύνθεση. Γι' αυτό ζητάμε να σταματήσουν οι διακρίσεις. Ζητούμε και γι' αυτό υποστήριζω την κυρία Λούνιτσεκ διότι ζητεί την ίση μεταχείριση ώστε να έχουν αυτοί οι άνθρωποι μια φυσιολογική ζωή το πολύ απλό του να μπορεί κανείς να ζει όπως του αρέσει και να μην χρειάζεται να παίρνει άδεια από κανέναν. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Η έκθεση θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου και την ευχαριστώ πολύ την κυρία Λούνα. Συνεχίσουμε τον αγώνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα κανένας δεν είναι υπέρ ε, των διακρίσεων νομίζω όλοι μας είμαστε υπέρ της ισότητας. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τις λεγόμενες θετικές ε, διαδικασίες, που τόσο ή άλλως διακρίσεις, είναι άρα παράδεκτες. Ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να ε, επιτρέψουμε στους ε, ΛΟΑΔ ιδιαίτερα δικαιώματα, συγκεκριμένα δικαιώματα. Η ισότιμη μεταχείριση αφορά όλους χωρίς καμία διάκριση. Ούτε προς τη μία κατεύθυνση θετική, ούτε προς την αρνητική. Αυτή η έκθεση ούτως ή άλλως παραβιάζει ε, κατάφορα τα εθνικά δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία. Ε, και ζητάτε μας επιβάλλετε την αμοιβαία αναγνώριση των ε, γάμων των ομοφιλοφίλων. Ε, όπως έχει πειωθεί πολλές φορές, ο γάμος είναι γάμος μεταξύ δύο ανθρώπων διαφορετικού φίλου με σκοπό την διαιώνιση του, του είδους. Όσοι είναι κατά των διακρίσεων, ε, θέλω αύριο να ψηφίσουν ε, την εναλλακτική πρόταση ε, του EFD, που θέλει να εξασφαλίσει τα δικαιώματα όλων, όχι μόνο των ομοφιλοφίλων. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να προωθεί στο Κοινοβούλιο. Η συνάδελφος Μέτσολα. Grazie. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην ε, κοινωνία ότι οι διακρίσεις βάρος των ΛΟΑΔ είναι απαράδεκτες. Είχαμε την ευκαιρία και την τον προηγούμενο μήνα να συζητήσουμε και με την κυρία Λούνατσεκ ε, να συμμετάσχουμε στις ε, συζητήσεις οι οποίες καταλήγουν σε αυτή την ισορροπημένη έκθεση. Έκθεση σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας. Έκθεση η οποία δεν αντιβαίνει στο δικαίωμα ενός κράτους μέλους να ρυθμίσει με βάση τις αρμοδιότητες που του ανήκουν. Θα σας εξηγήσω λοιπόν τι δεν κάνει η έκθεση. Δεν εισάγει νέα νομοθεσία. Ούτε μία χώρα δεν θα είναι υποχρεωμένη να θεσπίσει νομοθεσία που θα αλλάζει τις διατάξεις σχετικέ με την οικογένεια. Δεν θα αλλάξει τίποτα σε σχέση με την προσωπική κατάσταση των πολιτών. Δεν θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ζούμε τη ζωή μας στην κάθε χώρα. Αλλά θα ανοίξει το δρόμο η έκθεση αυτή για μια ποιοτική ζωή για όλους. Υπάρχουν κάποιες ειδήσει ε, ότι υπάρχουν διακρίσεις ει βάρος των ΛΟΑΔ όλο και πιο συχνέ. Γι' αυτό καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες με ένα οδικό χάρτη για την προστασία της γενετήσης ελευθερίας, της ίσης μεταχείρισης και καλό του πάντε να υπερψηφίσουν την έκθεση. Μπορσελίνο. She's Thompson. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή συνεργασία βασίζεται στην ελευθερία, τη δημοκρατία και την ισότητα και τον αλληλοσεβασμό για όλους. Ε, Παρ' όλα αυτά, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι ομοφιλόφιλοι στην Ευρώπη υφίστανται παρενοχλήσεις στον στο χώρο εργασία και αλλού. Ένα τέταρτο από αυτούς το 25% έχουν δεχτεί και δημόσιες ε, επιθέσεις. Είναι ώρα λοιπόν η Κομισιόν και το Συμβούλιο να αναλάβουν την ευθύνη τους για ε, την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων. Δέκα φορές έχουμε ζητήσει μια ε, συνολική σφαιρική νομοθεσία για την καταπολέμηση της ομοφοβίας στην Ευρώπη. Θέλω η Κομισιόν να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη ε, επί ενός νέου προγράμματος δράσης με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Η Κομισιόν θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα συμμορφωθούν επίσης με την ισχύουσα νομοθεσία και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο αύριο θα στηρίξει τις βασικές ε, αρχές, τις θεμελιώδεις αρχές. Η Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτή τη συζήτηση πήραν διάφοροι το λόγο και όλοι μίλησαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένας χώρος ελευθερίας, ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων. Αυτές είναι οι ιδέες μας, αυτές είναι οι σκέψεις μας. Όλοι πιστεύουν μάλλον ότι πρέπει να είναι έτσι. Αν κοιτάξουμε όμως την πραγματικότητα, βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους πολίτες διαφόρων κρατών μελών. Δεν είναι αλήθεια λοιπόν ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας άνοιξε το δρόμο για να καταπολεμήσουμε, κατά τον, να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις. Κοιτάξτε τις γυναίκες που δουλεύουν σε, σε εργοστάσια πολυεθνικών. Ε, κοιτάξτε ένα άτομο το οποίο δουλεύει στη Γερμανία σε εργοστάσιο και στη χώρα μου. Ε, στη χώρα μου θα κερδίσει 250 ευρώ, στη Γερμανία ή σε αντίστοιχες χώρες ε, δεκαπλάσια και θα είναι και καλύτερα προστατευμένο. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει, αυτή τη διάκριση πρέπει να καταπολεμήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και οι άλλοι υποβουλευτές, έχω κατακλειστεί από ε, ηλεκτρονικά μηνύματα που ισχυρίζονται ότι η έκθεση αυτή αποτελεί προσβολή της ελευθερίας του λόγου, γιατί καταδικάζει την ομοφοβία. Πολύ ηρωνικό όλο αυτό, πολύ παράδοξο, διότι αυτή τη στιγμή ακριβώς στην Ιρλανδία έχουμε μεγάλη λογοκρισία από τον ε, δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό εις βάρος του Ρόνι ο οποίος ήθελε να καταδικάσει ε, την ομοφοβία και μάλιστα καταδικάζονται και σε πρόστιμα πολλών χιλιάδων ευρώ ε, όσοι ε, μιλούν κατά της ομοφοβίας. Η όρτη λοιπόν, ο δημόσιος τηλεοπτικός σταθμό, είναι στα χέρια των συντηρητικών εκείνων που δεν θέλουν να αφήσουν ισότιμη μεταχείριση στο γάμο. Όταν ο Τζον Waters λέει ότι είναι ένα είδος σάτυρας ο γάμος των ομοφιλοφίλων, πρόκειται για ομοφοβία. Όταν η Μπρίντα O'Brien λέει ότι πρέπει η ισότητα να ειστερεί σε σχέση με το κοινό καλό, Πάλι ομοφοβία είναι. Και όταν έχουμε Ινστιτούτο στην Ιρλανδία το οποίο ε, αναπτύσσει υλοποιήσει εκστρατεία κατά του γάμου των, ομοφοβ, των ομοφιλοφίλων προπάλληλε η ομοφοβία είναι και εγώ θα παραλάβω τα λόγια του Ρόνιου Νίλ ότι πρέπει να ξεκουμπιστούν από τη ζωή μα αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κοινωνία μας έχει βασιστεί στις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι πολίτες της δικής μου χώρας ε, κοινωνούν αυτές τις αξίες και ε, ζουν και εργάζονται με αλλοσεβασμό και ταυτόχρονα σέβονται και την ελευθερία και τη δημοκρατία. Ε, είναι περήφανοι για τις ρίζες τους και τις παραδόσεις τους. Δεν αισθάνονται ότι κάνουν διακρίσεις εναντίον κανενός. Δεν είναι ομοφοβικοί. Γι' αυτό λόγο, κυρία Λούνατσεκ, πιστεύω ότι η έκθεση σας δεν μας αφορά. Το πρόβλημα δεν μας αφορά. Η έκθεση αυτή δεν μας αφορά. Κύριε Πρόεδρε, ως χριστιανοδημοκράτης φυσικά θέλω το σεβασμό της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων. Δεν θα πρέπει να ανεχόμαστε την ομοφοβία. Όταν ακούω όμως τον Ισπανό συνάδελφο να επικρίνει το ε, δημοψήφισμα για το γάμο στην Κροατία όπου το ένα τρίτο των ανθρώπων υπερψήφισε αυτή το συνταγματικό ορισμό του γάμου. Ε, Διερωτώ με θέλουμε να προστατεύσουμε τις ατομικές ελευθερίες ή να ξεκινήσουμε ιδεολογικούς πολέμους πριν τις ευρωεκλογέ. Γιατί μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν πρόκειται να αλλάξετε τα συντάγματα και συνταγματική, το συνταγματικό ορισμό του γάμου στην Κροατία αλλά ούτω ή άλλω δεν απειλεί το δικαίωμα κανενός. Τέλος θέλω να σα υπενθυμίσω ότι ακόμα και ο Πάπας Φραγκίσκος ε, υποστήριξε αυτόν τον ορισμό του γάμου. Και ακόμα και περιοδικά ε, γκέι τον ε, ανακήρυξαν τον άνθρωπο της χρονιάς. αλλά δεν πρέπει να συζητάμε τέτοια θέματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εμείς έχουμε κατακλειστεί από email που λένε ότι θέλουμε να δώσουμε και άλλα δικαιώματα στα άτομα ΛΟΑΔΑ. Η έκθεση αυτή δεν θέλει επιπλέον δικαιώματα, απλώς να, τους, να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, γιατί υφίστανται διακρίσεις οι άνθρωποι αυτοί καθημερινά στη ζωή τους. Πολλοί ε, υφίστανται και φυσική βία και μόνο μία, ε, ε, το ένα στα δεκάτομα καταγγέλει αυτά τα αδικήματα στην αστυνομία. Αυτό είναι απαράδεκτο για την κοινωνία μα. Είναι καθήκον μα να εξασφαλίσουμε την ισότητα για όλους τους πολίτες, ε, για την κοινότητα, την οικογένεια στα σχολεία κτλ. Στην Κροατία ε, το τα προγράμματα που προωθούνται σε αυτήν την κατεύθυνση ε, ήταν πολύ καλά και τα άτομα ενημερώνονται για τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών κοινωτές τους, έτσι μου είπαν. Όμως πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Ο, ο Επίτροπος Άντορ τώρα θα πάρει το λόγο. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Λούνατσεκ για την ε, σφαιρική της αυτή έκθεση. Η ομοφοβία ε, πλήττει την ε, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν συμβαδίζει με τις αρχές ε, και τις αξίες ε, στις οποίες ε, δράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν γνωρίζει τα προβλήματα των ατόμων ΛΟΑΔ ε, στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των διακρίσεων της βίας και του εκφοβισμού και επαναλαμβάνει ότι είναι προσιλωμένη στην καταπολέμηση αυτών των διακρίσεων στο όριο των αρμοδιοτήτων της. Παρ' όλα αυτά η βασική ευθύνη βαρύνει τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κομισιόν είναι υπέρ ενώ μια προσέγγιση με στόχους και για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ε, αυτή θα δώσει επίσης ε, παροχή ε, νομικής ασφάλειας, ασφάλειας δικαίου, ε, προστασίας των θεμάτων και επαναλαμβάνω ότι τέτοιου είδους στόχοι θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί. Η Κομισιόν ε, παρακολουθεί την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη, ε, όπως για παράδειγμα την οδηγία ε, απασχόλησης, την οδηγία για τα θύματα ποινικών αδικημάτων κλπ. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τα συμφέροντα των ατόμων Έτσι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Επιπλέον, πρόταση για οδηγία ή μεταχείρισης. Ε, εμείς ε, επιμένουμε στην διεύθυνση του ε, πεδίου εφαρμογή ε, σε όλα τα άτομα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 19 ε, της συνθήκης, για παράδειγμα, ε, ε του σεξουαλικού προσανατολισμού του χώρα εργασία αλλά και στην εκπαίδευση, στην κοινωνική προστασία κλπ. Ε, επίσης, για την ισότητα, η Κομισιόν συνεργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια για να στηρίξουμε τον αγώνα τους ε, στην καταπολέμηση των διακρίσεων εντίον των ΛΟΑΤΑ. Έχουμε δώσει χρηματική ενίσχυση, δημοσιεύσεις ε, και καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών. Επίσης, χρηματοδοτούμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις που υποστηρίζουν τα ίσα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤ και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον. Η έλλειψη ε, πρόσβαση σε ε, υγειονομικέ υπηρεσίε και σε μέτρα πρόληψης πολύ συχνά δημιουργεί στίγμα και διακρίσει, και μάλιστα πολλές φορές οδηγάει ε, και σε ανισότητες σε θέματα υγείας. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα με τις βέλτιστες πρακτικές. Στην Ευρωπαϊκή Έκθεση για δράση στο θέμα της υγεία και του, και του εργασιακού περιβάλλοντος θέλουμε τα άτομα ΛΟΑΔ επίσης να μπουν και στη μέση διάταξη του εθνούς, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ε, ε επίσης, ε, δηλαδή εκεί θέλουμε ε, αυτά τα άτομα να μην θεωρούνται ε, γιατί αυτή τη στιγμή ταξινομούνται, η κατάστασή του ταξινομείται ως ασθένεια. Θα συνεχίσουμε να καταπολεμούμε την ομοφοβία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και θα ε, συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε υπέρ της ισότητας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι για την ε, συνεχή σας ε, στήριξη στις προσπάθειές μας να προωθήσουμε την ισότητα. Συγχαίρω ξανά την εισηγήτρια. Thank you very much, Commissioner. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο. Η έκθεση Λούνατσεκ ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που αφορά στην έκθεση του κυρίου Ροσφόρ με θέμα εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και θέλω πρώτα να παρακαλέσω τον εισηγητή να πάρει το λόγο.